θα έχουμε λοιπόν μια ακρόαση όπως προβλέπετε και είναι εθιμικό στην Επιτροπή μας. Βλέπω πολλούς συναδέλφους οι οποίοι ήδη έχουν ζητήσει να λάβουν το λόγο. Θα ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία. Ο κύριος Μπρόινιγκς έχει καταρχήν την ευκαιρία να κάνει μια εισαγωγική παρέμβαση 10 λεπτών και μετά θα έχουμε διαδικασία επιτραπέζιας αντισφαίρησης με τη συμμετοχή των συναδέλφων οι οποίοι μπορούν να θέτουν ερωτήματα, ένα λεπτό για ερώτηση, δύο λεπτά για απάντηση και μπορεί να γίνει και μια συμπληρωματική ερώτηση για 40 δευτερόλεπτα και ο κύριος Μπρόνινς θα έχει ένα λεπτό για να απαντήσει. Κύριε Μπρόνιξ, εάν είσαστε έτοιμος, μπορούμε να σας δώσουμε κατευθείαν τον λόγο και να χρησιμοποιήσουμε υποφελώς τον χρόνο μας. Παρακαλώ. Thank you, uh, Mr. Chairman, esteemed members of the European... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη μου τιμή και με ικανοποίηση βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας σήμερα για να κάνουμε αυτή τη σύντομη ανταλλαγή απόψεων για τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Πριν να απαντήσω στα ερωτήματά σας, θα με τις ευκαιρίες, όπως είπε και ο Πρόεδρος, να σας παρουσιαστώ και να παρουσιάσω και ορισμένα στρατηγικά στοιχεία που αφορούν ε, αυτή την αρχή και μετά θα περάσουμε στον γύρο έρωτα απαντήσεων. Πρώτα απ' όλα, δύο λόγια για μένα. Βασικός ε, θεματικός τομέας ε, εμπειρίας ε, ήταν αυτός της έρευνας σε ό,τι αφορά ε, τις πολιτικές επιστήμες και στη θεωρία, αλλά περισσότερο ακόμα στην πράξη, σε σχέση με την έρευνα ε, βασισμένη ε, στην πολιτική για την ε, I4 ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένη της αξιολόγηση πολιτικών, παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων, εξελίξει ό,τι φορά την μεθοδολογία και τις μακροχρόνιες, τη μακροχρόνια διαμόρφωση πολιτικής. Η εμπειρία μου συνδέεται με διαφορετικά επίπεδα πολιτική. Σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε μελετήσει τη Φλάνδρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά και την έρευνα στα κράτη-μέλη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο όσα και στις διαδικασίες ε, παγκόσμιας ε, περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Τα τελευταία πέντε χρόνια είχα δημοσιεύσει σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση και έτσι έχω μια σε βάθος γνώση θεωρώ για το πώς ε, λειτουργούν αυτές οι περιβαλλοντικές πολιτικές και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τοποθετείται ως ε, φορέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, πέραν της ακαδημαϊκής μου έρευνας, συμμετείχα σε πληθώρα πολιτικών διαδικασιών, ε, σε διοικητικά συμβούλια, γνωμοδοτικά συμβούλια, αλλά και σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και φορείς ε, επιχειρηματικούς, είτε δημόσιους, είτε ιδιωτικούς, είτε και σε συμπρέξεις των δύο για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Ε, και σε ό,τι αφορά την βιώσιμη διαχείριση υλικών, Μπορώ εν γέννη να πω ότι εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα μεταξύ πολιτικής και πράξης, που είναι και ο ρόλος ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Σε ό,τι φορά την εμπειρία μου ε, στα ζητήματα ε, management, από το 1996 αφορούμε σε αυτό το τομέα και αυτή τη στιγμή ηγούμε το μεγαλύτερο Ινστιτούτο ε, τέτοιας πολιτικής στο Βέλγιο με τη προπολογισμό 6 εκατομμυρίων ευρώ και ο Γενικός Διευθυντής είμαι υπεύθυνο και για τον, για τον στρατηγικό προσανατολισμό, τη χρηματοδότηση και τις ε, σχέσεις με τα συναφή δίκτυα ενδιαφερομένων μερών και με τις διάφορες προεκτάσεις που έχει αυτή η θέση. Έχω ζήσει και εργαστεί σε διάφορες χώρες, ε, στις ΗΠΑ, στις κάτω χώρες ε, και έχω εκπονήσει έρευνα σε πολλές ε, χώρες, είμαι και γλώσσος, όπως βλέπετε τουλάχιστον τα αγγλικά καλά τα μιλάω, αλλά και άλλες γλώσσες. Και έχω πολύ καλές επαγγελματικές σχέσεις με Αμερικανούς και Κινέζους συναδέλφους σε ζητήματα που άπτονται του EEA. Από πλευράς ε, προσωπικότητας ε, είμαι υπέρ της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος σε όλο μου το επαγγελματικό βίο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ε, Βεβαίως και συμμερίζομαι το όραμα του e ε, σε ό,τι αφορά την εύρωστη αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι ο EA θα πρέπει να παράσχει αντικειμενικές αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες και να αποτελεί ε, διασύνδεση μεταξύ ε, διαφόρων διαφόρων μερών και ευρύτερα στην κοινωνία ακόμα αν θέλετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους ε, στόχους και προκλήσεις, έχω εντοπίσει τέσσερις, τη διατήρηση ε, της ποιότητας αλλά και ενίσχυση των ε, δραστηριοτήτων του EA γιατί έχει πολύ καλό ιστορικό αυτή η αρχή σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητές της αλλά απαιτείται συνεχιζόμενη προσοχή προς αυτά τα κύρια και βασικά καθήκοντα για να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο ποιότητας ε, παροχής πληροφοριών. Δεύτερον, η στήριξη των μακροχρόνιων και θεμελιωδών στατικικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αυτές τις ε, μεγάλες ε, αλλαγές. Το 2050 πλέον έχει γίνει το επόμενο αύριο σε πολλούς πολιτικούς ε, τομεί σε άλλους το 2030 είναι ο, ο πολιτικός ορίζοντας ε, σε ό,τι αφορά τι ε, τις πρωτοβουλίε πρωτοβουλίες για την ε, ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για την χαμηλότερη κατανάλωση άνθρακα. Είναι σημαντικό λοιπόν εμεί να προσπα... καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε αυτέ τι προκλήσει, απαντώντα στα εξή ερωτήματα. Ποια είναι η βάση γνώσεων που απαιτείται για να υπάρξει κατάλληλη χρηστή διακυβέρνηση σε τέτοια ζητήματα και τι είδου παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων απαιτείται. Μετά, ε, ε, η προσοχή που δίνουμε στην κοινωνιακή πτυχή αυτών των ε, μεταβάσεων, γιατί βεβαίως θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρη την κοινωνία. Και έτσι η δημιουργία μιας γνωσιακής βάσης που συνδέεται με ε, τους ε, κοινωνικούς φορείς εκτός ε, του στενού πολιτικού πλαισίου είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αυτή η προσέγγιση ευθυγραμμίζεται και με τις αναδυόμενες πρακτικές της κοινωνικής εκμάθησης σε ό,τι αφορά τη παραγωγή και διάδοση της γνώσης. Και βεβαίως οι συνδέσεις με τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά προγράμματα ε, είναι κύριο σημείο του προγραμματός μας. Το πρόγραμμα 2020, Ευζοία 2020, Living Well, μαζί και με το 7ο EAP, εστιάζεται ακριβώς ε, στο ζήτημα της ε, χαμηλής κατανάλωσης άνθρακας και της υγιούς ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών, που έχει μεταφερθεί και σε συγκεκριμένους στόχους. Ε, κάποια από αυτά είναι σημεία εστίαση για τον EA όπως η υλοποίηση, η πολιτική συνοχή, η συνοχή μάλλον στην πολιτική μας, αλλά και νέοι ε, στόχοι σε ό,τι φορά το αστικό ε, περιβάλλον και όχι μόνο, και η διασύνδεση, στενή διασύνδεση με τους ε, στόχους και τη διαδικασία ε, αυτών των μεταβάσεων που ανέφερα προηγουμένω. Είναι βεβαίω εξαιρετικά σημαντική η συνεργασία με τα ενδιαφέρομενα μέρη. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σημαντικό σημείο εστίαση, γιατί εκεί εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή και οι εμπειρογνώμονε που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και με τα χαράς μπορώ να πω ότι ε, για το επόμενο πολιετές ε, στρατηγικό πρόγραμμα του ΕΕ, τα πέντε, το πεντετές αυτό πλαίσιο, μέχρι να ενημερώσω ότι θα υπάρξουν δύο συνεδριάσεις, το Μάρτιο και το Μάιο, για να ενημερωθώ και εγώ με το τι συμβαίνει. Ευρύτερα τώρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν άμεσες διασυνδέσεις με το Κοινοβούλιο, το, την Επιτροπή και άλλα ε, συναφή σώματα και εταίρους για να διασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός μας ε, θα παράσχει ε, κατάλληλο έργο. Για τις σχέσεις μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχιστεί αυτή η παράδοση των ε, άμεσων και επικοδηματικών σχέσεων με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή συγκεκριμένα, όχι μόνο για τεχνικούς ή θεσμικούς λόγους, αλλά κατά τη γνώμη μου, γιατί και ως, προσωπικά ως δημοκράτης Πιστεύω πραγματικά στην ε, δημόσια επίβλεψη των πολιτικών διαδικασιών. Γι' αυτό βασιστείτε, μπορείτε να βασιστείτε στη δέσμευσή μου, ε, στις πολιτικές της δημοκρατικής διακυβέρνησης και με τα χαράς ε, να εμφανιστώ ενώπιόν σας ανατακτά χρονικά διαστήματα για να συζητήσουμε μαζί τις προτεραιότητες. Τώρα, μερικά ακόμα στοιχεία Κατανοώ ακόμα βεβαίως ότι υπάρχουν προκλήσεις ε, που, ε, που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουν επιπτώσεις και στον EEA, συζητήσεις που αφορούν τον προπολογισμό. Ε, επίσης η περιβαλλοντική πολιτική και πολιτική οικονομική διακυβέρνηση, ο ευρύτερος διάλογος για τον ρόλο ε, του οργανισμού και άλλα στοιχεία. Σίγουρα κατά τη διάρκεια των ερωταπαντήσεων κάποια από αυτά τα ζητήματα θα τεθούν. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ τιμή μου να εγούμε ενό τέτοιου οργανισμού ε, που έχει χέρι μια, μιας τόσο καλής φήμης ε, και σας εγγυούμε ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε το απαιτούμενο επίπεδο αριστείας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπρούινγκς για την εισαγωγική σας παρέμβαση και ξεκινούμε τώρα τη συζήτηση και θα δώσω καταρχήν το λόγο στους συντονιστές. Ξεκινώ με τον Ρίχαρτ Ζέιντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον διοριστέντα διευθυντή της ε, EEA. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πορεία που έχετε ακολουθήσει και ως επιστήμονας αλλά και ως εμπλεκόμενος στην τεχνολογική εξέλιξη η οποία προχωρά με έναν τρόπο ο οποίος είναι εκθετικός αλλά βυσικά ελοχεύει και πολλούς κινδύνους για το περιβάλλον και εμεί θεωρούμε ότι ο Ευρωπαϊκό Φορέα Περιβάλλοντο είναι ο κεντρικό φορέα ο οποίο πρέπει να επιληθεί των θεμάτων του περιβάλλοντο και να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα αυτή τη τεχνολογική εξέλιξη και να μα δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτέ τι εξέλιξει. Όπως ξέρετε, κύριε καθηγητά, υπάρχει η αρχή ήδη από τις ε, ευρωπαϊκές ε, συνθήκες και είχαμε και μια έκθεση τον περασμένο Δεκέμβριο με τίτλο από τον ε, Φορέα Περιβάλλοντος «Καθυστερημένα διδάγματα από έγκυρες προειδοποίησεις». Δηλαδή πρόκειται για το γεγονό ότι αν είχαν ελαιοποιηθεί εγκαίρω ορισμένε αποφάσει θα είχαν αποφευθεί πολλά προβλήματα. Παραδείγματο χάρη μπορεί να αναφερθεί το θέμα τη ε, υδροδότηση και των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί σε επίπεδο υγειονομικό με την υδροδότηση. Όλα αυτά βέβαια έχουν σημασία για την συγκεκριμένη σας εργασία και θα ήθελα να ξέρω πώς θα τα αντιμετωπίσετε. Δεύτερον, θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι δικές σας προσωπικές προτεραιότητες που έχετε θεσπίσει για την εργασία σας στον ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστώ κύριε Ζέμπερ που μείνατε πιστό στα δύο λεπτά. Ήταν ένα λεπτό βέβαια ο χρόνος ε, ερωτήσεως και για αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να μείνουν στο πλαίσιο του ενός λεπτού. Έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε κύριε Μπρούνικ. Στα πλαίσια των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων, η άποψη που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σωστή. Βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία. Πρώτο, όπως είπατε, είναι η αρχή της πρόληψης. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει το θέμα της αβεβαιότητας, της έλλειψης βεβαιότητας μάλλον, στην επιστήμη και βοηθάει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί με επιφυλακτικό τρόπο όπως και άλλοι πρωταγωνιστές στη διεθνή σκηνή. Δεύτερον, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μια ανάληψη ευθύνη σε επίπεδο συζήτησης δημόσιας πριν ληφθούν αποφάσεις. Σαν παράδειγμα συζήτηση για τα γενετικά τροποποιημένα. Υπάρχει μια συμμετοχή και διαβούλευση με το κοινό. Νομίζω επίσης ότι με τις νέες τεχνολογίες στην επιστήμη, σαν επιστήμον, θα πρέπει να περιμένει κανείς να είναι δεκτικός, ανοιχτός και σε σχέση με τις μελέτες επιπτώσεων και σε σχέση με τις αξιολογήσεις των κινδύνων. Το θέμα της επιστήμης λοιπόν συνδέεται με το ρόλο της, του Ιδρύματός μας Ταυτόχρονα όμως σεβόμαστε και την ιδέα της δημόσιας διαβούλευσης, συζήτησης για τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιάζουν ορισμένα θέματα για την κοινωνία και τον κόσμο. Τώρα σχετικά με τις γνώσεις που είναι διαθέσιμες Πράγματι υπήρξαν κάποιες προσπάθειες ε, για να υπάρξει μια προειδοποίηση. Το θέμα είναι αυτές τις ιδέες, τι τις κάνει η κοινωνία. Εμείς σαν Ινστιτούτο μπορούμε να παρέχουμε τις βέλτιστες δυνατές ιδέες με ένα θετικό όμως τρόπο και πιστικό τρόπο. Και πάλι πρέπει να σας παρακαλέσω, επειδή έχουμε πολλούς ομιλητές, να παραμείνετε πιστοί στους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα λεπτό κάνει κάθε ερώτηση και δύο λεπτά η απάντηση. Μετά έχει 45 λεπτά ο κάθε ομιλητής να θέσει συμπληρωματικό ερώτημα και η απάντησή σας δεν πρέπει να ξεπεράσει το ένα λεπτό. Επόμενος ομιλητής. Έχετε θέλετε κύριε Ζέμπερ θέλετε να θέσετε συμπληρωματικό ερώτημα. Όχι. Ο Γιώ Λάινεν για ένα λεπτό επίσης. Και από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Προφανώς το θέμα του Ευρωπαϊκού Φορέα Περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, για τις αναλύσεις που πρέπει να κάνουμε και οι δικές σας εμπειρογνωμοσύνες είναι και η βάση της νομοθεσίας και των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα σε εμά. Μαζί με άλλους συναδέλφους βρίσκομαι στην πλατφόρμα για μια Ευρώπη που, κάνει αποτεδοτική χρήση των φυσικών πόρων και ίσως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή η δραστηριότητά σας σε σχέση με τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Υπάρχει η προσέγγιση επί τη βάση του οικολογικού ίχνους, του footprint, ότι δηλαδή για όλα τα προϊόντα τα οποία παράγουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το ίχνος που αφήνει στο περιβάλλον και ποια είναι η διαδικασία του κύκλου ζωής τους. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν αυτό το θέμα στην, ε, στον φορέα σας, κύριε Μπρένιγκς. και το θέμα της αποδοτικότητας της ενέργειας είναι κάτι που συνδέεται με τα συστήματα παραγωγής και τα συστήματα κατανάλωσης των προϊόντων αυτών. Ταυτόχρονα και η αποδοτική χρήση των πηγών από πλευράς της Ένωσης είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την μεθοδολογία που ακολουθούμε για να ενημερωθούμε σωστά για το εάν ένα προϊόν είναι φιλικό ή όχι ε, με το περιβάλλον, αν είναι αποδοτικός ενεργειακά. Και εδώ μπαίνει η ιδέα του ίχνους του οικολογικού σε επίπεδο σε μικρό επίπεδο θα έλεγα του προϊόντος προσπαθούμε να κάνουμε μία ανάλυση του κύκλου ζωής του συγκεκριμένου προϊόντος και μία από τις προτεραιότητες του Ινστιτούτου μας αφορά τις κατηγορίες προϊόντων και θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των ευρύτερων στόχων πολιτικής που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρόπος που συνδεόμεθα λοιπόν και εξετάζουμε τα συγκεκριμένα προϊόντα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός θα πρέπει να εξετάζουμε τα προϊόντα και τις γραμμές παραγωγής και τις γραμμές κατανάλωσης οι οποίες είναι συγκεκριμένες, απτές και ορατές. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα πάντα και με τους πάντες. Απαιτείται να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους τομείς σαν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Ευχαριστώ. Υπάρχει συμπληρωματικό ερώτημα, κύριε Λάινεν. Ναι. Αναφερθήκατε στο 7ο πρόγραμμα δράση, με το οποίο θα πρέπει να επιληφθούμε και εμείς του χρόνου. Υπάρχει, υπάρχουν οι κλασικές προκλήσεις και οι νέες προκλήσεις. Οι νέες προκλήσεις είναι οι αβεβαιότητες για τη δημόσια υγεία, το φαινόμενο κοκτέιλ με την ε, δράση πολλών ουσιών, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, όλες αυτές οι ουσίες για τις οποίες δεν έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις. Είναι αυτό ένα από τα κεντρικά σημεία της ε, ενασχόλησής σας. Ένα λεπτό κύριε Μπρένιξ. Είναι πράγματι ένα θέμα το οποίο είναι κεντρικό στο έργο του φορέα περιβάλλοντος. Η σύνδεση μεταξύ υγείας και διάβρωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και επίσης το θέμα της χρήσης των νέων υλικών που μπορούν να έχουν επιπτώσει στην ανθρώπινη υγεία είναι μία από τις εννέα προτεραιότητες στο πρόγραμμα για το περιβάλλον της, Ευρωπαϊ... Ε, του Φορέα Περιβάλλοντος και γι' αυτό θα είναι θέματα τα οποία θα εμπλέκονται και στο πρόγραμμά μας. Όταν μιλάμε για νανοτεχνολογία και νέες τεχνολογίες αυτού του είδους, σας παραπέμπω στο πρώτο ερώτημα, <clears throat> όπου υπάρχει μια σαφή σύνδεση με την αρχή της πρόληψης και την ανάγκη να έχουμε εδρεωμένα επιστημονικά δεδομένα για να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα. Και υπάρχει πολλή αβεβαιότητα για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Γκεμπράντη για ένα λεπτό έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Γκρένιξ για την παρουσία του εδώ σήμερα ω ε, εκπρόσωπο ε, του EA. Έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Το ένα αφορά το μέλλον του οργανισμού σας. Ε, αν δούμε και τι συμβαίνει στις ΗΠΑ όπου υπάρχει αυτός ο οργανισμός ε, περιβαλλοντικής προστασίας, έχει πολύ περισσότερα καθήκοντα από ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Μιλάμε για κατευθύνσεις, για ε, επιθεωρήσεις και αυτή είναι και χείλος φτέρνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Ε, ποια είναι η θέση σας προς αυτό. Το δεύτερο ερώτημά μου αφορά τη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ως εισηγητής πολλές φορές αξιοποίησα τις γνώσεις που μας παρήχε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν συμβαίνει αρκετά συχνά, δυστυχώς. Αυτό τον τεράστιο πλούτο γνώσεων που ε, κατέχει ο οργανισμός σας, πώς ακριβώς θα το ε, διαθέσετε σε μεγαλύτερο κόμμα βαθμό στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα. Πρώτα απ' όλα για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ως ε, περιβαλλοντικού επόπτη στην Ευρώπη. Εφόσον υπάρχει ένα μεγάλο ε, χάσμα υλοποίηση σε κάποιες από τις περιβαλλοντικές πολιτικές, ε, η ιδέα αυτού του επιθεωρητή του επόπτη είναι χρήσιμη. Όμως πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τον πραγματικό ρόλο ε, της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή δεν ε, είμαι εκ πρώτης όψης υπέρ τη συμπερίληψη αυτού του στοιχείου στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Περιβάλλοντος, γιατί θα πρέπει ενδεχομένως να αναδιατυπωθεί η αποστολή και ε, ο στόχος ε, του οργανισμού. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός οργανισμός με διαφορετικές αρμοδιότητες που να αναλάβει κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συνάδει με τον τρέχοντα ρόλο του οργανισμού μας. Αυτό αφορά και την οικοδόμηση δυναμικού. Για το, αν, γίνει, αν γίνει ο οργανισμός μας ένας χωροφύλακας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα συμμορφώνεται και με τον πρώτο μας και πρωταρχικό μας ρόλο. Αυτή η έννοια έχει σχέση με την ε, συζήτηση για την υλοποίηση, όμως θα πρέπει πραγματικά να εξετάσουμε ποιος είναι και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σε αυτό το πλαίσιο. Το δεύτερο ερώτημά σα αφορούσε τον μεγάλο πλούτο γνώσεων στον EEA και κατά πόσο θα ενισχυθεί αυτός ο δεσμός ε, με το Κοινοβούλιο. Να απαντήσω συντομία ότι ε, αυτό εντάσσεται στο διάλογο για το επόμενο, επόμενο πενταετές πρόγραμμα και έτσι στους επόμενους μήνες ε, θα λάβετε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει συμπληρωματική ερώτηση. Η Σάτου χάσει τώρα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κανείς δεν ανέφερε προηγουμένως την ε, προκάτοχό σας, τη Τζάκη Μακλέη. Θα ήθελα να έχω τη δική σας άποψη <clears throat> για το ποιο τμήμα της εργασίας της, ιδίω τα θέματα αυτά, όπου ξεκίνησε νέες κατευθύνσεις στην, ε, στον Ευρωπαϊκό Φορέα Περιβάλλοντα, περιβάλλοντος, ποιους τομείς θέλετε να προωθήσετε εσείς και πού θα αλλάξετε κατεύθυνση. Ο Ρίχαρτ Σέμπερ αναφέρθηκε και σε αυτή την έκθεση για, τις, ε, για τα καθυστερημένα διδάγματα από έγκαιρες προειδοποίησεις που είναι μια θαραλέα έκθεση για τον τρόπο που εφαρμόζονται οι αποφάσεις, η λαμβάνονται υπόψη προειδοποίηση. Θα ήθελα να ξέρω εάν είσαστε διατεθειμένος να συνεχίσετε με ένα τέτοιο προορατικό και θαραλέο τρόπο στην προσπάθεια να δίδετε εγκαίρως τα στοιχεία αυτά σας στους λήπτες αποφάσεων. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Να πω ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών το EA, ο οργανισμός αυτός, έχει αναπτυχθεί πολύ. χαρακτηρίζεται από ένα πολλαπλασιασμό δραστηριοτήτων, μεθοδολογιών και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλεται εν πολλής και στην σοβαρότητα και την δράση και την καινοτόμο ικανότητα που επέδειξε η προκάτοχός μου. Είναι σαφές ότι αυτή η δυνατότητα πρόβλεψης είναι κάτι το σημαντικό εφόσον θέλουμε να παραμείνουμε σαν ένα όργανο το οποίο εσείς οι ίδιοι θέλετε να είμαστε. Νομίζω λοιπόν ότι το τελευταίο κομμάτι των τελευταίων δεκαετών εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ θετικό. Προφανώς και πρέπει να παίξουμε κάποιο ρόλο εφόσον θέλουμε να συνεισφέρουμε στην καινοτομία και την σωστή πολιτική χάραξη στην Ένωση. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Εγώ θα ξεκινήσω την 1η Ιουνίου. Δεν έχω πλήρη ενημέρωση για τα θέματα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αυτή τη στιγμή εξελίσσονται ε, στον οργανισμό. Θα προτιμούσα λοιπόν να μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τα έργα της Jacqueline Maclay Πάντως έχω την ένδειξη ε, ότι ακριβώς αυτά που έκανε είναι αυτό που πρέπει να είναι η υπηρεσία και αυτά θα δώσουν τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει η συγκεκριμένη οργάνωση. Κοιτάξτε από τα καθυστερημένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης εσείς γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο έρχεται σε επαφή η επιστήμη με την πολιτική. Εσείς σαν επιστήμον, ποιες πιστεύετε ε, ότι είναι οι περιβαλλοντικές απειλές που δεν έχουν γίνει ακόμα κατανοητές από τους πολιτικούς και οι οποίες πιθανώς να συμπεριληφθούν σε αντίστοιχες εκθέσεις σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα. Νομίζω ότι τα βασικά της γνώσης που δεν έχει εκτιμηθεί δεόντως από τους πολιτικούς και αυτό είναι κάτι που ξεπερνά και το δικό μας έργο, είναι κάτι το ευρύτερο γιατί μου θέσατε το ερώτημα ως επιστήμονα. Αν δείτε την κατάσταση της έκθεσης για το περιβάλλον και της ε, με καθυστέρηση ε, εκθέσεις έγκαιρης προειδοποίησης και την έκθεση εν πάση περιπτώσει για το περιβάλλον στην οποία παίζουμε κάποιο ρόλο είναι σαφές ότι η κατάσταση του πλανήτη ε, χειροτερεύει. Η βιοπικιλότητα ε, έχει αρχίσει και απομειούται ε, κλιματολογικές αλλαγές σημαντικές, ε, τα δάση ε, δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά, ο ρόλος τους, η παρουσία τους, οι ωκεανοί το ίδιο που βρίσκονται υπό απειλή και απαιτείται να δώσουμε περισσότερη προσοχή. Η Άννα Ρόσπαχ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα οποία λέτε βρίσκονται πολύ κοντά στα ερωτήματα που ήθελα να θέσω. Μιλάμε πολλέ φορέ για, την για τι ανανεώσιμε ενέργειε στην Επιτροπή μα. Μία από τι κύριε προκλήσει για την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια θα είναι η έλλειψη πόρων, φυσικών πόρων. Εάν μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε τα σκουπίδια και να τα ανακυκλώνουμε για παραγωγή ενέργεια, αυτό θα μπορούσε να λύνει και το πρόβλημά μα με τα, τα σκουπίδια. Μία από τι κύριε προκλήσει στον τομέα του περιβάλλοντο είναι και η ποσότητα πλαστικών που βρίσκονται στην επιφάνεια και στο βάθος της θάλασσας. Αυτό έχει αρνητικό αποτέλεσμα για το περιβάλλον, σκοτώνει τα ψάρια. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε την έμφαση στην ανακύκλωση ορισμένων μορφών αποβλήτων, όπως είναι τα πλαστικά, από συσκευασίες κτλ. Πώς θα είναι η προτεραιότητά σε αυτό λοιπόν. Δύο λεπτά λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα δεν θεωρώ ότι οφείλω εγώ να τα αντιμετωπίσω γιατί δεν είμαι εγώ υπεύθυνο για τη χάραξη πολιτικής. Υπάρχει όμως μια βάση γνώσεων που είναι απαραίτητη για να μπορέσουν και οι υπεύθυνοι να χαράξουν την πολιτική τους. Όμως η αλλαγή στην νοοτροπία ε, από την ανακύκλωση των απορριμμάτων ε, σε μία άλλη πιο βελτιωμένη πολιτική ε, που είναι θεμελιώδης και για το μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό πρότυπο για την ενεργειακή απόδοση. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, να δείτε την πηγή των απορριμμάτων. Το καλύτερο είναι να αντιμετωπίσουμε το, και να επιλύσουμε το πρόβλημα εκεί, στην πηγή του. Είπατε, ας πούμε, για τα πλαστικά που βρίσκονται στη θάλασσα. Κατέληξαν εκεί γιατί ε, κάποιος τα πέταξε στη θάλασσα από κάπου αλλού. και ο EA ε, στο, στην 7η πρόταση, στην πρόταση για το 7ο ε, πρόγραμμα δράσης έχει συμπεριλάβει ε, προτάσεις που το τέτοιων ζητημάτων. Πολλά, πολλά λοιπόν μπορούν να γίνουν και επί της ουσίας. Πώς δηλαδή περνάμε από αυτό τον κύκλο ζωής που στο τέλος έχουμε ένα πόρημα προς ένα πιο κυκλικό σύστημα αντιμετώπισης και διαχείρισης των πόρων, όπου μπορεί δηλαδή αυτό το παλιό απόρριμα να χρησιμοποιηθεί και δεύτερον ε, την ευρύτερη πολιτική. Αυτά λοιπόν είναι η βάση της απάντησής μου. Και για δύο αυτά τα στοιχεία ο EEA έχει παράσχει γνώση ε, προς τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών. Συμπληρωματικό ερώτημα, κύριε Ρόσπαχ. πολύ σύντομα. Θεωρείτε ότι αυτό το θέμα είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό δηλαδή για σας να μεταβιβάσετε αυτές τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας στους ευρωβουλευτές και ε, στους ευρωπαίους πολίτες. Ναι, βεβαίως και είναι σημαντικό να μεταβιβάζονται αυτές οι πληροφορίες γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ε, συζήτηση της, της ε, κατάλληλης διαχείρισης των πόρων ε, και ε, σε ό,τι αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Βεβαίω και υπάρχουν περιφέρειες που έχουν περισσότερα να κάνουν από άλλες και οι ίδιες οι εκθέσεις θα συμπεριλαμβάνουν τέτοια στοιχεία. Σε αντίστοιχε εκθέσει λοιπόν αναφέρεται ποια κρατημέλη έχουν ε, περισσότερες ε, δράσει να αναλάβουν σε σχέση με άλλε. Έχουμε κλείσει λοιπόν τον πρώτο γύρο ερωτήσεων από την πλευρά των συντονιστών. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων και θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Χιούμπνερ για ένα λεπτό. χωρίς μικρόφωνο. Sorry. The micro is not working. Το μικρόφωνο σας δεν δουλεύει. Please try another micro. Okay. Okay. Okay. Now. Okay. Sorry. Witam pana bardzo serdecznie i już trzymam Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω εδώ. Και εγώ εύχομαι ό,τι καλύτερο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είπατε ότι η επιστήμη δεν γνωρίζει σύνορα. Και ιδιαίτερα σε μια ενωμένη Ευρώπη η δήλωσή σας ήταν εξαιρετική και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Έχετε ήδη μέχρι τώρα συνεργαστεί επίσης και με ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Εφόσον λοιπόν γνωρίζετε την κατάσταση, πώς βλέπετε τα πράγματα. Θα μπορέσετε να συνεργαστείτε μαζί τους ε, και να διευρύνετε τις μορφές προστασίας του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, λέει ο κύριος Μπρούνιξ. Πράγματι, ο κόσμος της επιστήμης και μάλιστα κάτω από την αιγίδα της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο ε, διευρύνεται συνεχώς, βελτιώνεται και το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα θα δώσει ακόμα μεγαλύτερα κίνητρα και χαιρετίζω εδώ τα νέα ευρωπαϊκά δίκτυα που θα δημιουργηθούν με το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει συνεργασία και με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και με ερευνητικά κέντρα και δημόσια. Έχω εργαστεί μαζί τους, όχι όμως σε διευρυμένη βάση, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας γυτνίασης των νομοθεσιών σαν παράδειγμα είχα διδάξει λίγο στη Ρουμανία και με συναδέλφους από την Τσεχία, την Πολωνία, την Ουγγαρία. Έχω κάποια εμπειρία λοιπόν, χωρίς όμως να θεωρώ αυτό εμπειρογνώμονα για τα δίκτυα της ε, Ανατολικής Ευρώπης ε, για το περιβάλλον. Η υπηρεσία όμως έχει στενές σχέσεις, έχει ένα καλό δίκτυο, ε, συνεργάστηκε με τις χώρες αυτές και στην προκαταρκτική περίοδο πριν την ένταξη και συνεχίζεται μετά. Συνειδητοποιώ επίσης ότι πολλές φορές υπάρχει απόσταση που οφείλουμε να καλύψουμε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια. Θα πρέπει να γίνει άλλωστε εν μέρη και στις παλιότερες χώρες, το, η οργάνωσή μας λοιπόν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλα τα κράτη-μέλη και ξέρετε ότι έχουμε και την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων μας και στις χώρες γειτονίας, ε, οπότε και εκεί θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής. Συμπληρωματική ερώτηση. Πρόσφατα κατηγορήθηκε η υπηρεσία σας γύρω από θέματα διαφάνειας. Έχετε κάποιες προτάσεις από πλευρά σας να κάνετε έτσι ώστε να μην αμφισβητηθεί η διαφάνεια στους τρόπους λειτουργίας σας. Κοιτάξτε, γενικά έχω την αίσθηση ότι η διαφάνεια είναι η βάση της εμπιστοσύνης. Και η εμπιστοσύνη τι είναι. Είναι η βάση της σωστής δημοκρατικής λειτουργίας. Εκτιμώ λοιπόν σε βάθος την διαφάνεια. Από την άλλη δεν γνωρίζω καμία άλλη οργάνωση σαν τη δική μας η οποία να έχει τόσο ξεκάθαρους και αυστηρούς κανόνες στον τομέα της διαφάνειας, στον τομέα της σύμπτωσης και σύγκρουσης συμφερόντων κτλ. Το θέμα είναι λοιπόν να σεβόμεθα τους κανόνες οι οποίοι είναι ενισχύ. Δεύτερον, και κάτι το λιγότερο επίσημο θεσμικό αν θέλετε, και που φαίνεται στα πλαίσια της συζήτησης που ανοίγουμε για όλα αυτά θέματα με όλους τους άλλους ενδιαφερομένους και η Διαχειριστική Επιτροπή, το Διαχειριστικό Συμβούλιο της EEA ΕΕ κάποια από τα θέματα αυτά θα τα θεωρήσει κατά προτεραιότητα θέματα και θα τα αντιμετωπίσει. Ο κύριος Βιτόριο πρώτη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την εμπειρία την οποία εσείς ε, αντιπροσωπεύετε, εκφράζετε και συνεισφέρατε στην υπηρεσία αυτή. Να θέσω κάποιες ερωτήσεις πολιτικής περισσότερο. Αν και αυτό δεν είναι σίγουρα το βασικό κέντρο ενδιαφέροντος της υπηρεσίας. Η υπηρεσία αυτή καλείται να είναι σύμβουλος της Επιτροπής, σύμβουλος του Κοινοβουλίου εγώ ασχολούμαι ιδιαίτερα με την υπερθέρμανση του κλίματος και την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να κάνουμε μια επιπλέον προσπάθεια για μια νέα πολιτική η οποία θα μας επιτρέψει να στρέψουμε την προσοχή μας με μεγαλύτερη συνένεση σε παγκόσμιο επίπεδο για το πρόβλημα αυτό. Εσείς τι προτείνετε και τι θα προτείνετε στους επιτρόπους σας. Βεβαίω και συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Πρώτον για την ε, υπερθέρμανση ως ε, συνολικό ζήτημα, αλλά και αυτή την ε, μακροχρόνια διαδικασία για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Τα χρονικά σημεία του 2015 και του 2020 ως νέος ορίζοντας είναι συμφωνίας μπορεί να σας φαίνονται μακρινά, αλλά είναι πολύ κοντά. Υπάρχει λοιπόν προσπάθεια ανάληψη ηγετικού ρόλου σε πολλά από αυτά τα ζητήματα πολιτικής. Είναι σίγουρα η πιο φιλόδοξη ομάδα ε, χωρών που έχει δεσμευθεί σε κάποιες ε, αρχές πολιτικής. Κανένας άλλος ε, τέτοιο πυρήνα χωρών ε, δεν το έχει πράξει και μάλιστα ο πρόεδρος Ομπάμα προσφάτως ε, ανέφερε ότι πραγματικά θέλει να αναλάβει δράση για την υπερθέμαση του πλανήτη αλλά όπω ξέρετε χρειάζεται δύο τρίτα, πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία για να συνυπογράψει μια διεθνή σύμβαση. 67 γερουσιαστές λοιπόν χρειάζεται και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Αυτό λοιπόν αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Μετά, γιατί στην Κίνα κάποιοι θεωρούν ότι Υπάρχει ε, ταχύτατη αλλαγή στην οτροπία του κόσμου και πολύ πιθανό αυτό να συμβαίνει ε, και θεωρούν ότι αλλάζει και η κατεύθυνση σε τα τελευταία χρόνια και το 2006 είδαμε αυτό με συγκεκριμένε πολιτικές αποφάσεις ε, σε ό,τι αφορά τι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Παράλληλα όμως σε πολιτικό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία. Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ε, σε συμμαχίες που αφορούν χώρες ε, του παραδείγματος 1 και εκτός. Συμπληρωματική ερώτηση. Ε, η προσαρμογή στις κλιματολογικές αλλαγές είναι κάτι το οποίο έχει πολύ θα αποκριβεί. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω η υπηρεσία να μου πείτε πώς θα θέσει το θέμα αυτό και πως θα σταθεί απέναντι στο πρόβλημα με πολύ περισσότερο αποφασιστικό τρόπο. Ο κύριος Μπρούνιξ. Ήδη επενδύουμε πολύ προσπάθεια στην προσαρμογή και στο μετριασμό των αποτελεσμάτων της ε, κλιματικής αλλαγής. Μια έκθεση πριν από την διάσκεψη της Δόχα μίλησε για το χάσμα, το μεγάλο χάσμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της πραγματικότητας και των προβλέψεων. Υπήρξε λοιπόν αυτό το μήνυμα κινδύνου. Συνεχίζουμε λοιπόν την προσπάθειά μας για την προσαρμογή και το μετριασμό των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής, γιατί είναι φανερό ότι αντιμετωπίσουμε ήδη αλλαγές. Και η προσαρμογή θα είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον, που θα διαφέρει σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης. Επομένως χρειάζεται μια πιο διαφοροποιημένη αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γουτιέρες Κορτίνες, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Περισσότερα από όλα με απασχολεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλά κέντρα ερευνών στην Ευρώπη για τα θέματα αυτά και ο φορέας σας έχει γίνει ουσιαστικά ο φορέας που απαντάει τα ερωτήματα της Κομισιόν και δαπανά πάρα πολύ προσπάθεια, ενώ θα, θε, θα προτιμούσα να υπάρχει μια συστημική προσέγγιση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο συνεκτική πολιτική. Με εκπλήσει παραδείγματος χάρη το θέμα του, του, των υδάτων. Μιλάμε για όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την, ε, τον κύκλο του ύδατος, αλλά δεν μιλάμε καθόλου για την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στον κύκλο του ύδατος. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη εξάτμιση ύδατος από τη Μεσόγειο που το καλοκαίρι που το χειμώνα οδηγεί σε πλημμύρες. Δεν κάνουμε τίποτα για όλα αυτά. Η πολιτική μας θα πρέπει να έχει ένα παγκόσμιο χαρακτήρα. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο την γη, θα πρέπει να σκεφτούμε και την ατμόσφαιρα, τη βροχή, το κλίμα. Χρειάζεται μια πολιτική η οποία θα αντιμετωπίσει εν γέννη όλα αυτά τα προβλήματα. Και κυρίως μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για όλα αυτά τα ζητήματα. thank you. Ευχαριστώ για το ένα λεπτό, λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ και ο κύριος Μπρούνινγκ για τα ερωτήματα αυτά. Αν δούμε τα πιο εγκάρσια θέματα και την συστημική προσέγγιση, αυτό καταρχήν είναι κάτι το οποίο είναι η βάση της εργασίας του φορέα περιβάλλοντος τα επόμενα χρόνια. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αθεκτικότητα των οικοσυστημάτων σε μεγαλύτερη κλίμακα και ξέρω από την προετοιμασία που έχει λάβει η χώρα ότι αυτό θα παίξει ένα σημαντικό, ένα κεντρικό ρόλο στο έργο της EEA, του Φορέα Περιβάλλοντος. Δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω λοιπόν τη σημασία του ερωτήματός σας και την ανάγκη να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Συγχρόνως είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση γιατί προϋποθέτει ότι γνωρίζουμε όλες τις διασυνδέσεις και τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ διαφορών παραγόντων και για πάρα πολλά από αυτά τα θέματα παραμένει ακόμα πολύ έργο το οποίο πρέπει να γίνει, πολύ έρευνα η οποία πρέπει να γίνει και αυτό είναι ένα από τα καθήκοντα της EEA. Λέτε ότι δεν έχουμε μια αρκετά συνολική προσέγγιση και δεν θα πρέπει να παραμείνουμε μονάχα στην ε, εστίαση στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνω. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως για το προηγούμενο ερώτημα, η Ευρώπη είναι η μόνη ομάδα χωρών που έχει δεχτεί δεσμευτικά νομοθετήματα για την κλιματική αλλαγή και είναι έτοιμη να προχωρήσει σε διεθνές επίπεδο σαν μια ομάδα χωρών Επομένω, για μένα μια στεναρή ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι προπόθεση για να είμαστε ένα ισχυρό εταίρο σε δημόσιο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να παίξουμε λοιπόν και στα δύο γήπεδα εάν θέλουμε να διαδραματίσουμε αυτόν τον ρόλο, να είμαστε ηγέτες για τι ιδέε, τη γνώση και τι πολιτικέ. τα τελευταία 15 λεπτά, δευτερόλεπτα για τι πόλεις. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο έργο που πρέπει να γίνει για τα αστικά περιβάλλοντα και πιο καινοτόμα εργασία και σε επίπεδο Ευρώπης και παγκοσμίω. Yes. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το συμπληρωματικό ερώτημα, ήταν ήδη μέσα στο ερώτημά σας, λέει. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας, αλλά καλά λίγα τα στραβά μάτια, λέει ο πρόεδρος. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει πιο πολύ ενδιαφέρον τα μιλάμε για συστημικά θέματα. Εγώ βασίζομαι στη δική σας βοήθεια για να έχουμε μια πιο συστημική προσέγγιση. Όταν μιλάω για μια διεθνοποίηση, μιλάω για μια παγκοσμιοποίηση όλων αυτών των θεμάτων. Η Μεσόγειος δεν είναι μονάχα μια ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι ένα θέμα που εμπλέκει πάρα πολλούς. Πρέπει να δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο ποια είναι η σχέση μας με το κλίμα, όχι μονάχα τα θέματα του περιβάλλοντος, της θερμοκρασίας μάλλον, αλλά και άλλα ζητήματα. <laughs> Εντάξει. Πάλι είχαμε μια μικρή ε, υπέρβαση χρόνου, κύριε Μπρόινικ. Ναι, ναι, χαίρομαι που βλέπετε τη λάμψη στα μάτια μου όταν μιλάω για συστημικά θέματα. Είναι ουσιαστικά για την κατανόηση των μελλοντικών προκλήσεων τα συστημικά θέματα. Όταν μιλάτε για τη Μεσόγειο και πώς εγγράφεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για τη συνδέση με την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι οι κοινότητες γνώσης θα πρέπει να ξεπερνούν τα σύνορα και να έχουν μεγαλύτερη σχέση με το νότιο τμήμα του πλανήτη μας. Και χαίρομαι που ο ορίζον 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να παρακινήσει αυτή την παγκοσμιοποίηση των δικτύων γνώσης αλλά συγχρόνως συνδέεται και με την τοπική δυνατότητα δημιουργίας ικανότητας σε πολλές αυτές τις χώρες. Πολύ δύσκολο να έχει κανείς ένα σταθερό και ανθεκτικό σύστημα γνώσης όταν είναι ασθενείς οι θεσμοί. Και αυτό ξεπερνάει, ξεπερνάει το θέμα της γνώσης για το περιβάλλον. Ευχαριστώ, κυρία Κλάς. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Πίσω σας. Δεν με βλέπετε, δεν με βλέπετε. Εμείς θέλουμε πάντα όλο και περισσότερες εμπειρογνωμοσύνες σε επιστημονικό επίπεδο. Αλλά έχουμε και νέα προβλήματα όπως είναι αυτό των ενδοκρινικών διαταρακτών. Οι νέοι στόχοι απαιτούν και νέες προσπάθειες αξιολόγησης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς επιλέγετε τους επιστήμονες που διενεργούν μια έρευνα και πώς καθορίζετε και τα ερωτηματολόγια βάσει των οποίων γίνονται οι έρευνες αυτές. Είναι ρευστή η προβληματική με το περιβάλλον. Παραδείγματο χάρη, τα βιοκαύσιμα θεωρήθηκαν στην αρχή μια λύση για το, την κλιματική αλλαγή και την ανεξαρτησία της, ε, από την ενέργεια και τώρα φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα θετικέ λύσει. Πώ θεσπίζετε λοιπόν τι παραμέτρου με τι οποίε αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά ο Ευρωπαϊκό Φορέα Περιβάλλον και πώ μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι έχετε ε, αποτελέσματα τα οποία είναι αξιόπιστα σε επιστημονικό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Μπρόνιξ. Θεωρώ ότι η ερώτησή σας αφορά το τι είδους επιστήμονες και τι είδους επιστημονικές κοινότητες θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει. Κοιτάξτε, οι επιστήμονες ξεκινούν θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις και οι κατάλληλες ερωτήσεις προέρχονται εν μέρει από τις προηγούμενες γνώσεις, από την άλλη από κοινωνικές συζητήσεις, διαβουλεύσεις, και θα πρέπει κανείς να αναμίξει σωστά αυτές τις δύο μορφές για να διατυπώσει τις σωστές γεωστρατηγικές ερωτήσεις για το μέλλον. Αυτό είναι τμήμα της προσπάθειας που γίνεται για το επόμενο πενταετές πλάνο της υπηρεσίας μας. Αναφερθήκατε στα βιοκαύσιμα, σαν παράδειγμα θέματος επί του οποίου υπήρξε ε, διαμφισβήτητη επιστημονική πρόοδος και αμφισβήτηση των προηγούμενων γνώσεων πριν 10 χρόνια πολλοί θεώρησαν τα βιοκαύσιμα πανάκια ενώ σήμερα με το είδος της διαφάνειας της επιστημονικής η οποία χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση του θέματος τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα για την επιλογή των επιστημόνων και αν θα πρέπει να εξαρτώμεθα κάθε φορά από μία έκθεση, όχι, προφανώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να επωφεληθούμε από τα δίκτυα των επιστημόνων, όλο και περισσότερο διεθνή δίκτυα, όπως οι εκθέσεις του IPCC, η έκθεση GAP που κάναμε εμείς και πολλές άλλες διεθνείς εκθέσεις. Όλες αυτές είναι χρήσιμες και γι' αυτό θα πρέπει να, είμαστε, να σεβόμαστε τη διαφάνεια για την επιλογή των ομάδων των επιστημονικών οι οποίοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν τις πολιτικές μας αποφάσεις. Συμπληρωματικό ερώτημα, ναι, πάρα πολύ σύντομα. Όταν αξιολογείτε τις επιστημονικές μελέτες, παίζουν ρόλο και οι επιστημονικές ε, ερωτήσεις. Όταν μιλάμε για ένα, μια αναπολογισμό ε, κινδύνου σε σχέση με το περιβάλλον. Θα παίξουν ρόλο και επιστημονικά ερωτήματα. Αν πιστεύετε ότι τα θέματα του περιβάλλοντος συνδέονται με τα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης και τη διανομή του πλούτου και του κόστους και του ωφέλους στην κοινωνία μας, είναι λογικό να υπάρξει και οικονομική λογική η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη σε σχέση με την πολιτική του περιβάλλοντος. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε βεβαιασμένα τι είναι πολύ ακριβό ή τι είναι αυτό το οποίο εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα, δημιουργεί χάσματα ανταγωνιστικότητας. Τέτοιες, ε, τέτοιες χειρισμοί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πριν τους διατυπώσουμε αλλά σίγουρα υπάρχει αυτή η σύνδεση με την παραγωγή και τη διανομή και το κόστος και το όφελος. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά είναι και οικονομικά ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Η Κάριν ένα λεπτό. Να συνεχίσω λιγάκι με αυτά που είπε η κυρία Κλάς. Είσαστε ευρωπαϊκός φορέας, αλλά έχετε να αντιμετωπίσετε ευθύνες παγκόσμιου χαρακτήρα. Υπάρχει το θέμα της βιοποικιλότητας, παραδείγματος χάρη, και η χρήση της, το πρώτο θέμα, και το θέμα της βιομάζας και της χρήσης για παραγωγή καυσίμων. Ε, έχετε γνώση της ε, έρευνας της μελέτης αυτή που έγινε με την αίτηση της Κομισιόν για τα θέματα αυτά, θεωρείτε ότι μπορείτε να δεχτείτε αυτήν την ε, έκθεση ή χρειάζεται βελτιώσει και επίσης το δεύτερο της ε, έμεσης αλλαγής χρήσης γης και για το αν είναι απαραίτητο να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η σπορά σε ορισμένε περιπτώσεις. Και έχουμε δει παραδείγματα παραγωγικά την επίπτωση της αλλαγής των σπόρων που χρησιμοποιούνται στον πληθυσμό των μελισσών κτλ. Κύριε Μπρένιξ. Για το πρώτο ερώτημα για τη βιομάζα, όπως είπα, Ακόμα και πριν από πέντε χρόνια, πολλοί θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό λύση για το ενεργειακό μας πρόβλημα. Αλλά σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, δυσκολίες, προβλήματα και μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Μετά για την χρήση γης ε, και την αλλαγή στη χρήση γης ε, που συνδέεται και με τη γεωργία. Και αυτό προ... ξεπερνά μάλλον τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντο Ταυτόχρονα όμως εμείς ζητούμε μια καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε ε, μεγαλύτερες εμβέλειες ε, πολιτικές όπως είναι η κοινή πολιτική και αυτό συνδέεται με την ε, χρήση γης, ε, τα αποτελέσματα που θεωρούμε επιθυμητά ή όχι, και σα παραπέμπω σε τέτοιου είδου αιτήματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντο ε, για τα διατομιακά θέματα. Ε, για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, εγώ στηρίζω το ευρωπαϊκό σύστημα που βασίζεται στην αρχή της ε, πρόληψης, που είναι πιο αυστηρό σε σχέση με τις ΙΠΑ, την, τη Χιλή ή αλλού την προβολή και δημοσίευση των επιστημονικών δεδομένων, τη δυνατότητα δημόσιας συμμετοχής και μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Όμως, εδώ η ΕΦΣΑ βεβαίως και έχει τον ηγετικό ρόλο. Και παρακολουθεί αυτές τις διαδικασίες. Ως επιστήμον, και ως επιστημονικό, ε, επιστημονικός φορέας βέβαια και πρέπει να μείνουμε ανοιχτοί απέναντι σε τέτοιου είδους συστήματα. Η επιστημονική ορθοδοξία και ο δογματισμός δεν ε, μπορούν να ενταχθούν στο δικό μας πλαίσιο. Υπάρχει κάτι άλλο. Συμπληρωματικό ερώτημα ε, θεωρείτε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να αναλάβετε εσεί τα ίνια για θέματα όπω είναι αυτά που άπτονται και τη ασφάλεια των τροφίμων. Μα νομίζω ότι η κατανομή των ε, καθηκόντων μεταξύ των φορέων υπόκειται σε αποφάσει που έχουν ήδη ληφθεί. Η ΕΦΣΑ υπάρχει για να αντιμετωπίσει τα θέματα ασφάλεια τροφίμων και για την αντιμετώπιση όλων αυτών των διαδικασιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο, αλλά δεν πρέπει να είναι ένας ρόλος ο οποίος θα είναι γενικός. Αυτή τη στιγμή περιοριζόμαστε στο να δούμε τις πτυχές του περιβάλλοντος και έχουμε πάρει ήδη μια θέση για τα θέματα αυτά σε σχέση με την περαιτέρω ε, ολοκλήρωση των πολιτικών βάσει της ε, έκθεσης GAP. Υπάρχει ήδη λοιπόν η κατανομή ευθυνών. Αν αλλάξει αυτή μπορεί η EA ΕΕ να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο, αλλά αυτό είναι μια διαφορετική συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερνάντης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο α, ε, Διευθυντή, τον κύριο Μπρένεξ και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία. Θα ήθελα να σταθώ στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο προτείνεται από το Συμβούλιο. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη για αυτό το πλαίσιο για το διάστημα 2014-2020 σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και πώς θεωρείτε ότι πρέπει να δράσουμε για να πετύχουμε τους στόχους που αφορούν το περιβάλλον και που απορρέουν από τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και επίσης που προέρχονται από το πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 2014-2020. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι η δική σας θέση έναντι της πρότασης του Συμβουλίου και έναντι των στόχων που το Συμβουλίο και η Κομισιόν έχουν διατυπώσει. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να δράσουμε για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Η συζήτηση που γίνεται είναι πολιτική συζήτηση και εξάγεται αρκετές μέρες τώρα και στο Κοινοβούλιο. Η γνώμη πολλών από τους ευρωβουλευτές είναι διαφορετική από την γνώμη στο Συμβούλιο και, στο, και στην Επιτροπή. Εμείς λοιπόν σαν υπηρεσία θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα. Να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες και για τον δικό μας προϋπολογισμό. Όταν λέω αναμονή δεν εννοώ παθητική αναμονή, έχουμε επιχειρηματολογήσει προς την Επιτροπή, έχουμε πει ότι εφόσον μας θέλετε να κάνουμε τα συγκεκριμένα πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να έχουμε τα μέσα για να το πετύχουμε. Αν μικρύνει ο προπολογισμό, τότε θα πρέπει να επιλέξουμε κάποιες προτεραιότητες, να προσπαθήσουμε δηλαδή να βρούμε μια κάποια ελαστικότητα χωρίς όμως να διαρρήξουμε την ισορροπία μας. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτοί που θα είναι υπεύθυνοι για τα επόμενα πέντε χρόνια που θα ξεκινήσει η περίοδος αυτή τον Ιούνιο, οι περικοπές, οι περικοπές χρηματοδότησης να μην θίξουν τα βασικά προγράμματα της υπηρεσίας και αυτοί οι οποίοι ζητούν η υπηρεσία να αναλάβει περισσότερα έργο, περισσότερους στόχους και υπηρεσίες να το κάνουν αυτό στα πλαίσια ενός πνεύματος ρεαλισμού. Γιατί πάντα εργαζόμαστε στα πλαίσια ενός αρκετά περιορισμένου δημοσιονομικού πλαισίου. Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα που θα συζητήσω όταν αναλάβω μαζί με την ε, ε, ομάδα διαχείρισης στο Συμβούλιο το Διαχειριστικό. Συμπληρωματικό ερώτημα. Φέτος είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών και φανταζομαι ότι πολύ λίγοι πολίτες γνωρίζουν το φορέα σας και αυτά τα οποία πράτετε. Και αναρωτιέμαι σε αυτό το έτος των πολιτών πώς θα κάνετε πιο ορατό το έργο του φορέα σας και πώς θα μπορέσετε να, ε, να προσελκύσετε τους Ευρωπαίους πολίτες στο να κατανοήσουν και να προωθήσουν τους στόχους του περιβάλλοντος. Ίσως μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία απάντηση στα τελευταία χρόνια ο φορέας μας τα τελευταία 5 με 10 χρόνια έχει αναπτύξει ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας ώστε να πλησιάσει τους πολίτες και να κάνει γνωστή τη λειτουργία της περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Είναι λοιπόν ορατός ο φορέας μας και η ορατότητα αυτή είναι μία από τις προτεραιότητές, προτεραιότητές μας. Και μέλη του φορέα μας έχουν έρθει σε επαφή με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με κοινωνικούς εταίρους σε διάφορες συζητήσεις. Και ένα τμήμα της ε, συζήτησης πράγματι προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ε, ανησυχίες και τις ενασχολήσεις του στο επόμενο πενταετές σχέδιο. Αυτές οι επαφές λοιπόν θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο η επικοινωνία με τους πολίτες και η παροχή με έναν τρόπο που να είναι κατανοητό και σχετικό με την εμπλοκή του στην διαμόρφωση πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Παύλ Κόκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Θα ήθελα να επανέλθω στη σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και τη ΕΦΣΑ, γιατί πολλέ φορέ γίνεται λόγο για επικαλύψει. Ε, προσφάτως αναφερθήκαμε στα νεονικοτονοειδή και τους ενδοκρινικούς ε, διαταράκτες. Ε. υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών και θα θέλατε να βελτιωθεί αυτή. Νομίζω ότι, για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω και πολλά για τις σχέσεις μεταξύ ΕΦΣΑ και EEA. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ε, δεν ε, είχα τη δυνατότητα να το εξετάσω τους τελευταίους μήνες. Μου λείπουν λοιπόν ε, κάποιες γνώσεις αυτή τη στιγμή για να σας πω ακριβώς πώς έχουν αυτές οι επαφές και αν, αν θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις. Σε αδρέ γραμμέ θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και άλλων οργανισμών θα πρέπει να βασίζεται ε, πρώτον σε σαφή καθορισμό ε, και επιμερισμό των ε, αρμοδιοτήτων για να μην υπάρχουν επικαλύψει. Δεύτερον, να λειτουργούν συμπληρωματικά σε ό,τι αφορά τη γνώση, να συμπληρώνουν δηλαδή ο ένας τις ενέργειες του άλλου και φαντάζομαι ότι σε ορισμένα ζητήματα θα ήταν καλό να συσταθούν προγράμματα δράσης, δίωδη επικοινωνίας, ακόμα και εκθέσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό όμως είναι δυνατό. Για κάποια ζητήματα που συλλέγουμε πληροφορίες και γνώσεις, ίσως θα μπορούσε να υπάρχει λοιπόν ένας πιο δεδομένος τρόπος ανταλλαγής. Όμως, για να είμαι ειλικρινής και πάλι λέω ότι δεν γνωρίζω πώς έχουν οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και ΕΦΣΑ. Ευχαριστώ. Επερώτηση. Ναι. Η ΕΕ πέρσι δημοσίευσε μια τεχνική έκθεση και η Επιτροπή τώρα προετοιμάζει ε, νομοθετική ε, πρόταση. Ποια είναι η γνώμη σας? Για μια ακόμη φορά θα προσπαθήσω να είμαι ειλικρινής και να πω ότι δεν έχω συγκεκριμένες γνώσεις. Δεν μπορώ να κάνω κάποια δήλωση γι' αυτό. θα πρέπει να συνεχίσω το διάβασμα στις συγκεκριμένες εκθέσεις. Τρίτος και τελευταίος γύρος ερωτήσεων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μόρκουνάιτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρόνιγκς που είναι μαζί μας σήμερα και να θέσω μια ερώτηση σχετικά με τη Βαλτική. Όπως γνωρίζετε η Βαλτική είναι η πιο μολυσμένη θάλασσα στον κόσμο. Ε, ε, γνωρίζετε τους λόγους. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα με στόχο την μείωση των φωσφορούχων που έχουν πέσει στη θάλασσα θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να γίνει η οικολογία μας ή η γεωργια μας πιο οικολογική. Το θέμα βέβαια είναι ότι όλα αυτά ασχολούνται με το μέλλον, ενώ η μόλυνση είναι παρούσα σήμερα. Έχετε υπόψη σας αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί ήταν επαρκή ή ήταν έγκαιρα. Και αναφέρομαι εδώ στον αγωγό πετρελαίου Nord Stream Ακούσαμε ότι μετά από την κατασκευή αυτού του δικτύου έχει αυξηθεί η μόλυνση στην Βόρεια Θάλασσα. Κοιτάξτε, είπατε ότι η Βαλτική είναι από τις πιο μολυσμένες, αν όχι οι πιο μολυσμένη. Αυτό συνδέεται με την ιστορία της εκβιομηχάνησης αλλά και τις μορφές άσκησης της γεωργίας στην περιοχή. Για το αν επαρκούν τα μέτρα, προφανώς όχι δεν επαρκούν Απαιτείται περαιτέρω πρόοδος για την ποιότητα του περιβάλλοντος. Αυτό είναι προφανές. Τώρα για το τι είδου μέτρα μπορεί κανείς ρεαλιστικά να αναλάβει στην περιοχή το ταχύτερο δυνατόν, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει με πολιτικούς όρους σχετικά με τις αποδεκτές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν οι χώρες που περιβάλλουν τη Βόρεια Θάλασσα και οι κοινοτικές και οι βαλτικές και οι σχέσεις μας με την Ρωσία. Αυτό παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες γιατί εμείς σαν, ή σαν οργάνωση έχουμε επαφές και με το Σκανδιναβικό, στο το Βαλτικό Συμβούλιο Συνεργασίας Τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει όμως με την απαιτούμενη ταχύτητα και αυτό δεν αφορά μόνο τις βιομηχανικές ε, ε, σχέσεις αλλά και τις θεσμικές επαφές μας με την περιοχή. Προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς έχει σημασία, σε ποιο επίπεδο μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν θα πρέπει να θίξουμε την ανταγωνιστικότητα σαν παράδειγμα. Όλα αυτά συνδέονται με τα θέματα του περιβάλλοντος αλλά είναι σαφές οι αριθμοί, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μέτρα που πήραμε είναι ανεπαρκή και νέες παρεμβάσεις όπως ε, ε, ο αγωγός ε, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να ειδωθεί πριν ληφθούν οι αποφάσεις επί τη βάση των μελετών επιπτώσεων κυρίως. Μάλιστα, μία συμπληρωματική ερώτηση. όταν γίνει η, προτεραιότητα, Προεδρία Λιθουανική, η βασική της προτεραιότητα θα είναι η στρατηγική για τη Βαλτική. Και θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της περιοχής σε πολλούς τομείς και θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε θέματα που άπτονται της οικολογία. Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα καλύτερης εφαρμογής της στρατηγικής της Βαλτικής. Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε δηλαδή τις υπηρεσίες και τα όργανα να συνεργαστούν καλύτερα. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω ε, στα πλαίσια της άποψης που έχει η οργάνωσή μας. Εμείς συνεργαζόμαστε μέχρι τώρα σωστά και με την Προεδρία, οπότε ε, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα περιβαλλοντικά προγράμματα στα οποία αναφέρεται η Λιθουανία Ξέρω ότι προετοιμάζεται ε, και συνεργάζεται με τη Λιθουανία για τα θέματα αυτά. Δεύτερον, η βελτίωση της στρατηγικής για τη Βαλτική δεν είναι μία απλή απόφαση, δεν είναι μία επιλογή καν της EEA. ΕΕ. Νομίζω ότι αυτοί που θα αποφασίσουν να ενισχύσουν τη στρατηγική αυτή μπορεί να υπολογίζουν στην Ε.Ε. Ε, σαν γνώστης της κατάστασης και των δυνατοτήτων παρέμβασης και σε επίπεδο δημιουργίας δυνατοτήτων, κυκλοφορίας των πληροφοριών, παροχής επιστημονικών βάσεων, τεκμηρίωσης αποφάσεων, εκεί φυσικά θα συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Χάουκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρόινικ έχετε ηγηθεί δεξαμενών σκέψης και επιστημονικών Ινστιτούτων. Τώρα είσαστε επικεφαλής ενός φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως τμήμα της διοικητικής μηχανής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως εμπλέκεστε και στον προεπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολιετές και σε ετήσιο επίπεδο. Εμεί ξέρουμε ότι ο, ο προπολογισμό είναι ένα θέμα εξέχουσας πολιτικής σημασίας. Βλέπετε όμως ότι ούτε η Κομισιόν ούτε το Συμβούλιο παίρνουν στα σοβαρά αυτά τα οποία λένε. Λένε λόγια αλλά δεν τα εφαρμόζουν. Το ερώτημα μου τώρα το εξή. Με ποιο τρόπο θέλετε, τουλάχιστον στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματός σας, να εφαρμόσετε όλα αυτά τα μέτρα, να έρθετε σε επαφή με τους εταίρους σας μέσα στην διαδικασία του προϋπολογισμού και πώς θα συνεννοηθείτε με το Διοικητικό Συμβούλιο. Πώς θέλετε λοιπόν να πολιτικοποιηθούν ορισμένα θέματα ώστε έναντι των κρατών μελών να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πράγματι ένας τακτικός και επαρκής προϋπολογισμός για την EEA. Λέτε ότι δεν είσαστε λήπτης αποφάσεων, αλλά θα πρέπει αν θέλετε να έχετε ένα πραγματικό προϋπολογισμό να εμπλακείτε σε αυτές τις ερωτήσεις. Κύριε Μπρούνιξ. θα πρέπει να γίνω πολύ ισχυρό στρατηγικό συνήγορο για τον ρόλο ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντο και αυτό απαιτεί και προπολογισμό, χρηματοδότηση. Θεωρώ ότι ε, τα δύο κύρια στοιχεία που μπορεί να αξιοποιήσει ο EEA με τι διαπραγματεύσει ε, με όσου θα καθορίσουν τον προπολογισμό μα είναι η αναγκαιότητα του έργου που διεξάγει ο οργανισμός μας, γιατί κανένας άλλος δεν το κάνει, και η ποιότητα και το γεγονός ότι προκύπτουν και νέες ε, απαιτήσει. Και υπάρχει και ένα όριο ε, στην ε, αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Βεβαίως και θα προσπαθήσουμε εμείς να είμαστε πιο αποδοτικοί στο έργο μας, αλλά υπάρχει και ένα όριο σε αυτά. Τι κάνει λοιπόν ε, το Διοικητικό Συμβούλιο και πώς μπορούμε να το εμπλέξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει ε, να συμμετάσχει στα πιο στρατηγικά στοιχεία της λειτουργίας ε, του EA και αυτό έχει γίνει στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τις πιο σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή εκπονούμε το επόμενο πενταετές σχέδιο. Πρέπει να είναι σαφές και είναι σαφές ότι οι συζητήσεις επί είναι μια συνθήκη, μια συγκυρία που πρέπει να ληφθεί υπόψη και η τρέχουσα, η φυστάμενη ε, ηγεσία του ΙΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν επίγνωση του γεγονότο ότι θα πρέπει να λάβουν θέση εκεί και αυτή η θέση θα πρέπει να ε, μεταβιβαστεί στις Γενικές Διευθύνσεις και στο Συμβούλιο. Από εκεί πέρα είναι μια πολιτική απόφαση. Πάρα πολύ σύντομα στο διπλωματικό ερώτημα. 20 δευτερόλεπτα. Είσαστε έτοιμος επομένως. Όταν η Κομισιόν σας δίνει όλο και περισσότερα καθήκοντα κάποια στιγμή να ζητήσετε χρήματα ή αν δεν σας δίνουν τα απαραίτητα χρήματα να απορρίψετε την ανάληψη αυτών των αρμοδιοτήτων ή όχι. Τώρα, για να σας το πω πιο διπλωματικά, ε, Εάν μα ζητά κανεί περισσότερε αρμοδιότητε, αλλά δεν μα ε, δίνει μεγαλύτερο προπολογισμό, τότε θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητε. Ε, τα νέα καθήκοντα ίσω να αποτελέσουν ε, προτεραιότητε βεβαίω, αλλά πρέπει να τα επανεξετάσουμε όλα από την αρχή. Και πάλι όμω υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε στην επόμενη περίοδο. Μαργαρέτα Οκέν, øh. Ε, καλώς ήλθατε στην Κοπενχάγη, κύριε Μπρόνιξ. Πρέπει να συνηθίσετε και τα δανέζικα, γιατί αυτά θα ακούτε μέρα νύχτα στην Κοπενχάγη. Ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε καλή συνεργασία μαζί σας, όπως είχαμε με τη Ζακλίν Και όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι. Απαντούσατε ένα ερώτημα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και την ΕΦΣΑ. Και σχημάτισα την εντύπωση ότι είχατε την αρχή της ε, πρόληψης την οποία εφαρμόσατε ως επιστήμον στα θέματα αυτά. Η αρχή της πρόληψης όμως έχει να κάνει και με την προστασία του περιβάλλοντος και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι πρόβλημα για το περιβάλλον. Η αρχή της πρόληψης δεν σημαίνει ότι οι επιστήμονες θα πρέπει να κάνουν έρευνα. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς που έρχονται να μας πούν για το περιβάλλον και αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει ένα ανοιχτό πνεύμα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στη σύμβαση του όρχους υπάρχει και κάποια αμνία της απαραίτητης διαφάνειας Εντάξει, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Μπρονίξ. Τα δανέζικά μου αυτή τη στιγμή είναι πολύ ανεπαρκή. Αλλά θα πάρω ιδιωτικά μαθήματα, ιδιαίτερα μαθήματα για να βελτιώσω κάπως τα λίγα δανέζικα που ξέρω. Και δεύτερον, μιλήσατε για την καλή συνεργασία με την Jacqueline Μακλέιτ. Το είπα στην αρχή, όχι επειδή πρέπει να το κάνω εδώ, αλλά επειδή το λέω σοβαρά, θέλω να δημιουργήσω μια αντίστοιχη σχέση μαζί σας, όπως και η προκατοχός μου, για τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και την αρχή της πρόληψης. Σίγουρα είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Σίγουρα οι επιστήμονες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και έρχονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες όταν συζητούν τα θέματα αυτά και εξαρτάται η θέση τους από την προέλευση τους πολλές φορές και την προηγούμενη τους πορεία. Μια πρόσφατη έκθεση του ΦΑΟ που βασιζόταν σε επιστημονικές δημοσίευσεις ανέφερε τα υπέρ και τα κατά για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αβεβαιότητα για την τελική αξιολόγηση. Σε ορισμένου τομεί είναι πιο σαφή τα πράγματα, σε άλλου λιγότερο. Σαν φορέας διαχείριση τη γνώσης πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτό πνεύμα και κριτικό πνεύμα σε σχέση με τις γνώσεις οι οποίες ε, εμφανίζονται για τον τομέα αυτό, ακριβώς γιατί είναι ένα επίμαχο θέμα και η δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη. Επομένω, το να έχουμε σαφείς γνώσεις και να έχουμε μια πιο υγιεινή, λέει ο συζήτηση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξασφαλίσει η επιστήμη και η διαδραστική επιφάνεια μεταξύ επιστήμης και πολιτικής που είναι η EEA. Ευχαριστώ. Επτά δευτερόλεπτα για τη Μαργαρίτα. είσαστε πάρα πολύ σκληρό με αυτού που είναι από άλλε πολιτικέ ομάδε λέει στον πρόεδρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μου απάντησε ο κ. Μπρονίξ για αυτό που είπα για την σύμβαση του όρχου. Μιλάμε εδώ πέρα για την αρχή της πρόληψης σαν να είναι απλώς μια επιστημονική ιδέα και όχι ένας τρόπος αντιμετώπισης της υγείας και της φύσης. Και πάλι νομίζω ότι η βιοπικιλότητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της αρμοδιότητάς σας. Πρώτον, συνειδητοποιώ πλήρω ότι η αρχή τη πρόσληψη έχει σαν στόχο την προστασία του περιβάλλοντο, την προστασία τη υγεία και γι' αυτό και στηρίζω την αρχή αυτή και γι' αυτό στηρίζω και την ερμηνεία που δίδει η Ευρώπη σε αυτή. Και όχι την πιο φιλελεύθερη, αν θέλετε, ανάγνωσή τη, την οποία κάνουν διαφορετικοί εταίροι. Δεύτερον, γνωρίζω και την ε, σύμβαση του Όρχους, ε, γνωρίζω και τις πόλεις της Δανίας, και γνωρίζω τη σημασία που έχει η Σύμβαση του Όρχους στην δημιουργία του δικαιώματος για μια ξεκάθαρη συζήτηση για την βιοπικιλότητα και να υπάρξει και σωστή ενημέρωση των πολιτών της κοινωνίας. Είμαι υπέρ αυτού του είδους διαφάνειας ε, και δικαιώματος του κοινού να ενημερώνεται. Θα συμφωνήσω λοιπόν ε, με αυτό το οποίο υποβόσκει στην ερώτησή σας. Η σας ευχαριστώ. Το ερώτημά μου ακολουθεί το τελευταίο ερώτημα, αλλά με διαφορετική προσέγγιση, γιατί και εγώ ήθελα να μιλήσω για την αρχή της πρόληψης και την ανάλυση των κινδύνων. Ένας από τους κύριους στόχους της CEA ΕΕ είναι το να, παραθέτω, να δώσει έγκαιρα και σχετικά στοιχεία και αξιολογήσεις των στοιχείων που έχουμε και το γνώσεων και το περιβάλλον. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι οι αξιολογήσεις δεν βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου, αλλά μόνο στην αντίληψη των πιθανών κινδύνων, που είναι μια διαφορετική κατεύθυνση κατά τη δική μου άποψη, παρά, ε, παρόμοια. Αν, πάρουμε, αν αναλάβουμε δράση από τη βάση της αρχής της πρόληψης και των ενδεχόμενων κινδύνων, ίσως δεν λαμβάνουμε πάντα υπόψη τις ε, απρόβλεπτες συνέπειες των δράσεών μας. Γιατί αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε κάτι, εμπλέκονται άλλες ουσίες, γίνονται άλλες ενέργειες οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα για το περιβάλλον χωρίς να το έχουμε προβλέψει αυτό. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν και εγώ ένιωσα κάποια ανησυχία όταν διάβασα αυτή την έκθεση τα καθυστερημένα μηνύματα από έγκαιρε προειδοποίησεις στο κεφάλαιο περί υπάρχει εντύπωση ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία των επενδεδημένων συμφερόντων, βιομηχανικών κύκλων, μπλα μπλα κτλ. Δεν υπάρχει σαφή διατύπωση. Αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σα στάση για τα θέματα αυτά και αν είστε διατεθειμένοι να προχωρήσετε σε πραγματική, ε, σε πραγματική ανάλυση κινδύνων μέσω τη CEA. Πρώτον, όταν κάνει κανείς μία ανάλυση των κινδύνων και την αξιολόγησή τους, στα πλαίσια της διεθνούς φιλολογίας θα δει ότι υπάρχει μια συνένεση, ότι αυτό αποτελείται από δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το περισσότερο αντικειμενικό και το έτερο είναι υποκειμενικότερο. Πρώτον, η αντίληψη για το φαινόμενο είναι πολύ σημαντική και αφορά το μέγεθος του κινδύνου και τις πιθανές συνέπειες για την κοινωνία μπορεί να αποδεχθεί κανείς και να διαχειριστεί. Βλέπετε λοιπόν ότι και το αντικειμενικό κομμάτι και το υποκειμενικό είναι συστατικά απαραίτητα για την αξιολόγηση του κινδύνου και θα πρέπει να ισορροπούν μεταξύ τους. Θα συμφωνήσω επίσης ότι απρόβλεπτες συνέπειες πολιτικών θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε κάποιες διαδικασίες αξιολόγησης εκ των προτέρων. Εγώ έχω προσπαθήσει να εξετάσω μετερολογικά τις ε, πιθανόμενες σκοπούμενες ή μη σκοπούμενες συνέπειες πολιτικών και άσκησής τους στο περιβάλλον και ιδιαίτερα σε επίπεδο μετεωρολογικό. Ουσίες σαν παράδειγμα οι οποίες μπορεί να αντικαταστήσουν το όζον το οποίο συρρυκνούται. Υπάρχει σιγά σιγά επιστημονική γνώση για τα θέματα αυτά. Μεθοδολογικά λοιπόν, αυτή θα ήταν η απάντησή μου. σχετικά και για τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και την καθυστερημένη κυκλοφορία τους. Εγώ δεν έχω συνεισφέρει στην σύνταξη αυτών των εκθέσεων. Οι γνώμες που έχω είναι προκατηλημένες, προκαταλαμβάνω αν θέλετε τις, τα στοιχεία με βάση τις δικές μου προσωπικές απόψεις, ως εκ τούτου δεν είναι σωστό να κάνω σχόλιο. Κοιτάξτε, στο τελευταίο κομμάτι η απάντηση ήταν ενδιαφέρουσα, γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτά τα έγγραφα, εφόσον μείνετε στη θέση σας όσο και ο προκάτοχός σας, θα παραμείνουν και αυτά σε ισχύ για μία δεκαετία τουλάχιστον, οπότε διαρωτώ με αν θα διαφωνήσετε ε, με τα στοιχεία αυτά. Κοιτάξτε, εγώ δεν διαφωνώ με τίποτα σε αυτή τη φάση. Δεν είναι αυτός ο στόχος ε, της ακροάσεώς μου. Θα ήθελα όμως να ξεκαθαρίσω ότι υποστηρίζω τα συμπεράσματα της έκθεσης. Είναι συμπεράσματα τα οποία βασίζονται σε ένα μεγάλο όγκο γνώσης η οποία είναι καρπός του τι κέρδισε η επιστήμη από τις συζητήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και μέχρι τώρα. Έχω κάνει μια αντίστοιχη προσπάθεια σε μικρότερη κλίμακα για τη Φλάνδρα στο Βέλγιο. Νομίζω λοιπόν σαν όργανο οργανογνώσεις είναι υποχρέωσή μας να φέρουμε στην επικαιρότητα και την ιστορία των γνώσεων που είχαμε στο παρελθόν και τις συνέπειες της εφαρμογής τους. Ευχαριστώ. Έχουμε κλείσει λοιπόν του τρίτου και του τελευταίου γύρου ερωτήσεων απαντήσεων. Ο κύριος Μπρόνιξ έχει την δυνατότητα να, δώσει μια τελική, να κάνει μια τελική δήλωση πέντε λεπτών, εφόσον το επιθυμεί. Okay, well, I, I think I will keep it even shorter than... Λιγότερο ακόμα και από πέντε λεπτά θα μιλήσω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, ανοιχτές και ειλικρινείς σας ε, ερωτήσεις εδώ σε αυτό το γύρο ερωταπαντήσεων. Τα ερωτήματά σας περισσότερο αφορούσαν τις διαδικασίες, τη χρηματοδότηση, τα ενδιαφέρμενα μέρη ε, και το περιεχόμενο, το ρόλο του οργανισμού μας στο πλαίσιο των ευρύτερων περιβαλλοντικών πολιτικών. Για μένα αυτό καταδεικνύει και το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στην Επιτροπή σας για αυτά τα θέματα και τη στήριξη όμως που μας δείχνετε και βεβαίως θα την αξιοποιήσουμε για να συνεργαστούμε μαζί σας στο μέλλον. Και επαναλαμβάνω εδώ τη δέσμευσή μου απέναντι στην Επιτροπή σας. Ξέρω ότι είχατε εξαιρετικές σχέσεις με την Τζάκλ Μαγκλέιτ και σκοπεύω να συνεχίσω την παράδοση. Κατανοώ επίσης από αρκετά ερωτήματα ότι υπάρχει ζήτηση για να χρηστεί κοινοποίηση του έργου ε, του Οργανισμού Περιβάλλοντος, ε, πέραν και της ε, Επιτροπής εδώ. Αυτό σίγουρα εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσης του EEA και εγώ θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα προσωπικά. Αναφερθήκατε και σε ζητήματα ε, λογοδοσίας και διαφάνειας. Για μένα η διαφάνεια είναι η βάση της εμπιστοσύνης και η εμπιστοσύνη είναι η βάση της συνεργασίας. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε επί του περιεχομένου και πραγματικά είναι κάτι το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα. Από τη συζήτηση προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τις πιο καινοτόμες ε, επιστήμες και επιστημονικές εξελίξεις, ε, όπου υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα και ως επιστήμον μπορώ να σας πω ότι εξορισμού ε, όταν υπάρχουν αβεβαιότητες ε, πρέπει να γίνει να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες και να γίνουν πολλές εργασίες. Και αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, σε συνεργασία και με εσά και με το Συμβούλιο και την Επιτροπή κάποια από εσάς αναφέρθηκαν σε ζητήματα που υπερβαίνουν ε, τα όρια των μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, είτε είναι από τη Μεσόγειο, είτε από τη Βαλτική, είτε από αναπτυσσόμενες χώρες. Και στο παρελθόν ο ρόλος μας ήταν ε, ο ρόλος ενός ε, ε, ιδρύματος αναφοράς ε, για τέτοια ζητήματα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν αφορά δηλαδή μόνο στενά ε, αυτή την Επιτροπή, αλλά ευρύτερα και άλλους φορείς. Όπως ξέρετε, είμαστε, και λέω είμαστε παρόλο, παρότι δεν είμαι, είμαι ακόμα, δεν έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου, έχουμε εκπροσώπους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ε, και εκπονούμε το επόμενο ε, πρόγραμμα. Έχουμε δημοσιονομικούς περιορισμούς ε, και υπάρχει και πολιτική συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το προετοιμάζουμε, το προετοιμάζουν μάλλον οι υπάλληλοι με το πιο σοβαρό δυνατό τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει γνώση των ε, επίμαχων ζητημάτων και κατανοεί ότι είναι στρατηγική σημασία για το μέλλον αυτό το πρόγραμμα και ελπίζουμε ότι θα βγούμε πιο δυνατοί, με ένα πιο δυνατό ε, πρόγραμμα από αυτή τη διαδικασία, αλλά και ρεαλιστικό ταυτόχρονα που θα το επιτρέψει να διατηρήσει τον κεντρικό του ε, ρόλο και ελπίζω έτσι να αποτελέσουμε ένα ισχυρό εταίρο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και βεβαίω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία μαζί σα. Ευχαριστώ. Yeah, Θέλω σας ευχαριστήσω κύριε Μπρόνινς για τις απαντήσεις που μας δώσατε σήμερα, για την παρουσίασή σας και για το γεγονός ότι κάποια ερωτήματα είπατε ότι δεν μπορείτε να τα απαντήσετε τώρα αλλά θα προκύψουν από την εργασία μου στο μέλλον. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός φορέας, ο φορέας του περιβάλλοντος για μας, η EA, για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και όπως είπαν και ορισμένοι συνάδελφοι και εμείς βασιζόμαστε σε μια ενίσχυση της συνεργασίας μαζί σας γιατί σίγουρα μπορούν οι εκθέσεις μας να βελτιωθούν με την καλύτερη συνεργασία μαζί σας και με τη χρησιμοποίηση της εμπειρογνωμοσύνη σας, γιατί εμείς ως Κοινοβούλιο δεν έχουμε δική μας πηγή εμπειρογνωμοσύνης, αλλά είναι ένα κενό το οποίο μπορείτε εσείς ως EEA να το καλύψετε. Περνάμε τώρα στην συζήτηση μεταξύ συντονιστών για να μπορέσουμε να συντάξουμε μία επιστολή η οποία θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν διαβιβαστεί στους αποδέκτες της. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εύχομαι να έχουμε μια καλή συνεργασία στο μέλλον, μια στενή συνεργασία και προφανώς είσαστε πάντα ε, καλοδεχούμενος στην Επιτροπή μας όταν θέλετε. Έχουμε κλείσει λοιπόν την ημερησία διάταξη. Θέλω να χαιρετήσω και μια ομάδα επισκεπτών που ήδη είχα χαιρετήσει και χθε από την Γενική Διεύθυνση μετάφραση από το Λουξεμβούργο που ήρθαν εδώ 16 ασκούμενοι είσαστε το μέλλον της υπηρεσίας μετάφρασης και γενικά της εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σημαντική προφανώς για το έργο του Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι έχετε πάρει μια καλή εντύπωση από την εργασία του Κοινοβουλίου. Στις 5.30 λοιπόν θα λάβει χώρα η συνεδρία των συντονιστών και κλεισμένο των θυρών. Για το σημείο 16 έχω να κάνω μια ανακοίνωση 25 και 26 του μηνός θα συνεδριάσουμε το απόγευμα της 25ης από τις 3 το πρωί και το πρωί της 26ης έχουμε ψηφοφορίες και συνεχίσει των συζητήσεων. Κλείνει η συνεδρίασή μας και σας εύχομαι καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.